Ολοκληρώθηκε αυτό το στάδιο κυρίε και κύριοι. Έχω μία ανακοίνωση. Οι αρμόδιε αρχέ τη Κροατία ε, μου διαβίβασαν ένα μήνυμα για την άρση τη ασυλία του κυρίου Ιβαν Γιάκοφτσιφτ και βάσει του άρθρου 9 παράγραφο 1 του κανονισμού το αίτημα παραπέμπεται στην Επιτροπή Νομικών Θεμάτων.